Colleagues, meanwhile, we can adopt the agenda. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν έχω να σας κάνω ανακοινώσεις, αλλά μπορώ να σας κάνω μια αποσαφήνιση για το θέμα των προφορικών τροπολογιών, γιατί στη τελευταία συνεδρίασή μας είχαμε ένα, μια σύγχυση συστήνω σε όσους ε, ε, θέλουν προφορικές τροπολογίες πρώτον να το δείξουν καθαρά σηκώνοντας το χέρι τους, δεύτερον ότι ε, θα πρέπει να διαβαστεί η τροπολογία αυτή καθαρά από τον υποβάλλοντα την τροπολογία. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουν δηλαδή οι συνάδελφοι χωρίς να ξέρουν το κείμενο. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Προσπαθώ να κερδίσω και λίγο χρόνο, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, λέει ο Πρόεδρος. Yes, now we do the test, but... So, meanwhile we start with the test. Εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε πρώτα μία δοκιμή. Άρχεται η ψηφοφορία. Μου έπεσε και το σφυρί. Thank you very much. Oh. Still six colleagues to vote. Έχουμε ακόμα έξι συναδέλφους που δεν έχουν ψηφίσει. Ε, υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν ε, τις κάρτες τους μαζί τους. Ο Πάρτο Μπράιαν, ο Ρενάτο. Εντάξει. Μου λένε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η κάρτα του Μπράιαν και όπου να είναι θα φτάσει, δεν μπορώ να περιμένω άλλο όμως. Θα, σας, θα μετράμε τις ψήφους επιπλέον. Άλλη μία κάρτα. Μονάχα ένας ε, από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ε, λείπει, δηλαδή δεν έχει κάρτα. Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν να ψηφίσουμε τον ε, κανονισμό για το Money Market Fund. Είναι ένα πολύ σημαντικό νομοθετικό θέμα. Ψηφίζουμε την τροπολογία 224 υπέρ. Κατά. Ε, νομίζω ότι απερίφθη, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Απερίφθη. Τροπολογία 21 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 225 υπέρ κατά βλέπω ότι όλοι έχουν πλέον την κάρτα τους αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 22 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός α τμήμα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ε, κάναμε ένα λάθος. Στην σελίδα 4 αναφέρεται θα πρέπει να γράψουμε if rejected σε περίπτωση που ε, απορριφθεί, όχι if adopted σε περίπτωση που εγκριθεί. Επομένως, ε, βεβαίως, εδώ υπάρχει ένα λάθος τυπογραφικό. 261 υπέρ, κατά, αποχές, 264 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 262 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 265 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος επί της 265 Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 266 υπέρ. Κατά. Αποχές. <clears throat> Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 266, παρακαλώ. Για δέστε στο διπλανό μηχάνημα μήπως λειτουργεί. Πολύ ωραία. Vote is closed. Is rejected. Απερίφθη. 267 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση 267. Πέρας. Απερίφθη. 268 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 269 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά το αποτέλεσμα είναι πολύ σφιχτό. 269 <clears throat> ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται ψηφοφορία. Ακόμα δύο πρέπει να ψηφίσουν. Δεν θέλουν να ψηφίσουν, δεν πειράζει. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 271 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2,70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2,72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2,73 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 2,73 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 2.75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.77 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία 2.77. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβασμός H πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός I πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός J πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 339 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 340 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 340 άρχεται. Απερίφθη. Συμβιβασμός B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 375. 357 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 359 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, αλλά να το ελέγξουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την ε, τροπολογία 359. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 364. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται συμβιβασμός O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 397 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 398 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 398, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβασμός και η υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 422 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται αλλά φαντάζομαι ότι θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά βεβαίως άρχεται η ψηφοφορία Έχουμε μία ψήφο σοσιαλιστών παραπάνω. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. Τροπολογία 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 425 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 424 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται να κάνουμε τον έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν πρόσεξα καλά. Με ακούλπα. 4.24. Πέρας. Απερίφθη. 4.26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά να το τσεκάρουμε. Τροπολογία 426, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 428 υπέρ Παρατηρήσει εκτό μικροφώνου, δεν ακούν οι διερμηνείς. yeah. I, thought you could see it. Uh, 428. 428 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 430 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη συμβιβασμός π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 478 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 479 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 481 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 480 είναι ταυτόσιμη γιατί δεν το γράφει εδώ ωραία 482 λοιπόν υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. 482, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται. Απερίφθη. 485 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 484 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 486 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 486 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 487 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 489 ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 490 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 492 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβασμός D πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 410 συγγνώμη 5-10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4-96 τι είναι, είναι η ίδια με του εισηγητού. 4-96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5-12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός ή πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 3 Α, όχι, διορθώνει ο Πρόεδρος. Δεν υπάρχει τμήμα 3 και εδώ έχουμε ένα τυπογραφικό λάθος. Όχι if adopted, αλλά if rejected.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 Ε, τμήμα 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πηγαίνουμε λοιπόν στο συμβιβασμό V. σε τρία τμήματα επίσης πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ένα α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε στην τροπολογία 557, Αλέν Λαμασούρ και Αλέν Καντέκ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμός τι, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός γιου, Α, πάμε στη σελίδα 36 απευθείας. U, ε, τμήμα 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τμήμα 2, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός W, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 706. Πηγαίνουμε απευθείας. Λοιπόν, ε, ψηφίσαμε όχι την 78 αλλά μια, την άλλη τροπολογία η οποία είναι ταυτόσιμη, δεν έχει σημασία λοιπόν. Επομένως, συμβιβασμός G υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, συμβιβασμός X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 745 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 747 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 746 υπέρ, κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Επί της 746 άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. Τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 748 υπέρ κατά Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Τροπολογία 748 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 749 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 750 υπέρ τες απορρίπτεται. 751 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 753 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 752 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 752 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 754 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 754 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 755 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός S υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός Y για τον άρθρο 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ In favor, ε, είστε υπέρ ΕΛΚ, α, είστε κατά. Πώς, ποιοι είναι υπέρ του 98. Κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 98. Vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας απεριφθεί. Τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Τροπολογία 100, ναι, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική υπαλήθευση επί της τροπολογίας 100, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 102 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 102 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 103 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 103. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104 υπέρ κατά απορρίπτεται 105 υπέρ κατά Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά καλύτερα να το ξαναδούμε. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 105. Πέρας. Απερίφθη. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω τις ψήφους της Άλντε. Α, απερίφθη. Την απορρίπτεται. Ωραία, απερίφθη. τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 108 άρχεται η ψηφοφορία απερίφθη τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά καλύτερα να το δούμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 112 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 Φτάνουμε στην 118, οι άλλες έχουν καταπέσει, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός Z, πρώτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 2, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 3, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 129, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 130, υπέρ όχι, συγγνώμη, 131, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 132, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 133, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 134, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 135, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 ε, υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 138 άρχεται η ψηφοφορία. εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Όχι, πηγαίνουμε απευθείας στην τροπολογία 139 υπέρ κατά αποχές. Ε, δεν είμαι βέβαιος. Μάλλον όχι, εγκρίνεται, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 όχι αυτό καταπίπτει 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 146, γιατί ούτε οι 146 είναι όλες ε, ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές. Ε, τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ κατά ε, ψηφίζουμε. 147 κατά αποχές εγκρίνεται 148 κατά αποχές ε, απορρίπτεται ε, συμβιβασμός ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 155 υπέρ κατά εγκρίνεται Τροπολογία 158 υπέρ κατά αποχές ε, έλεγχος επί της 158 άρχεται εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Right, in favor, against... 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την 169 υπέρ, άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 170. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Επί της τροπολογίας 170 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία AC τμήμα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πηγαίνουμε στην τροπολογία 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2.11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2.12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. We 212 and we... 2.14. Ψηφίσαμε τη 2.12 και πάμε στη 2.14. 2.14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 19 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 2.15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 2.15 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Άρα πάμε στη 2.19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και επομένως θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 2.23, όχι ούτε την 2.23, ε, οι υπόλοιπε έχουν εκπέσει και επομένως διονομαστικής κλήσεως η τελική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. 34 ψήφοι υπέρ, 18 ψήφοι κατά, 5 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν με, ε, με απόλυτη πλειοψηφία. Τώρα να ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία επί του ψηφίσματος νομοθετικού περιεχομένου. Vote is closed. Πέρας. 35 ψήφοι υπέρ, 18 κατά, 3 αποχές. Η εισηγήτρια θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Για την επόμενη ψηφοφορία ήθελα να σας πω τα εξής. Εάν είμαστε υπέρ εδώ, ε, θα πάμε σε τριμερή διάλογο. Διαφορετικά, αν καταψηφίσουμε, θα περάσουμε από Οπότε ήθελα να καταλάβετε ακριβώς τι θα συμβεί σε κάθε περίπτωση ε, ψήφου. Η δική μα απόφαση ήταν να περάσουμε την Ολομέλεια του Απριλίου. Απλώ θα ήθελα η Προεδρία να ξεκαθαρίσει τι θα συμβεί εάν υπερψηφίσουμε ή καταψηφίσουμε. Δεν χρειάζεται να καταψηφίσουμε για να περάσουμε από την Ολομέλεια. Αυτό λέω εγώ. Σβέν, θα ήθελα, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, συνάδελφοι, να ακούσουμε προσεκτικά. Η έκθεση που έχω εδώ λέει πως το Συμβούλιο πραγματικά δεν είναι κοντά στη συμφωνία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην περάσουμε από την Ολομέλεια για το θέμα αυτό. Γιατί είδαμε ότι υπήρχαν κάποια πολύ στενά περιθώρια και πολύ μικρές διαφορές. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε η έκκληση σε όλους να περάσουμε από την Ολομέλεια, να ψηφίσουμε εκεί. Σβέν, ναι, αυτή είναι και η δική μας πρόταση και η πρόταση της ηγήτριας τότε εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα να περάσει το θέμα από την Ολομέλεια. Το δικό της ερώτημα στο οποίο εγώ αποφάσισα, απάντησα αρνητικά είναι για το αν για να περάσουμε από την Ολομέλεια πρέπει να καταψηφίσουμε την εντολή για τριμερή διάλογο. Και εγώ απαντώ πως δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν μπορούμε να ψηφίσουμε επί της πρότασης της ηγήτρες και να περάσουμε από Ολομέλεια. Λοιπόν, υπέρ. Χρειαζόμαστε ονομαστική ψηφοφορία. Αυτό είπα. The proposal of the rapporteur to go to the Ακούσατε τι είπε η συγκήτρια. Για περάσουμε από ολομέλεια. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Θέλετε ονομαστικά. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Για να περάσουμε από την Ολομέλεια. Να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Άρα έχουμε σχεδόν ομοφωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. say something? Uh, you have to use the Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, να ευχαριστήσω τους σκιώδες σίτες, να ευχαριστήσω τους βοηθούς, τη γραμματεία και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη σας, ε, για όλη σας τη βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolleginnen und Kollegen, ich wäre Ihnen dankbar, Sie würden gerade platzen. Οι συνάδελφοι θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν ήσυχα. Οι υπόλοιποι παρακαλώ καθίστε για... και σταματήστε επιτέλους την συζήτηση. Κούκου, ου, συνάδελφοι, ε, ευχαριστώ. Σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη. Δείκτες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, ως ε, συγκριτικοί δείκτες αξιολόγησης. Θα δώσω τον λόγο λοιπόν πρώτα απ' όλα συνάδελφο Φων Κόρα, Παρακαλώ. Χάουζεν, σχεδόν, σχεδόν καλά το είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχει συνεχιστεί σταθερά η δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα της ελευθερίας μας Και έχουμε τώρα τις πρώτες συμβιβαστικές τροπολογίες από τη Δευτέρα. Τις τελευταίες 15 μέρες είχαμε κάποιες ε, συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές και χαίρομαι που βλέπω πως ε, όλοι συμφωνούμε με αυτό το θέμα, ειδικά τώρα που το Συμβούλιο συμφώνησε με τη Γενική Προσέγγιση, πρέπει να βιαστούμε. Αναμένω τώρα την ε, συζήτηση για τις ε, προτινόμενες ε, συμβιβαστικές αυτές ε, τροπολογίες και την ανταλλαγή απόψεων με τους κοιόδης εισηγητές. Ευχαριστώ κόρα για το ΕΛΚ. Ο Λούντεκ Νίντερμαϊερ έχει πρώτο τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω την κόρα και την ομάδα της για τη φανταστική δουλειά που έχει κάνει και τα πράγματα πάνε μια χαρά κατά την ε, άποψή μου. Να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε δύο ζητήματα. Πρώτον, αναλογικότητα, ειδικά σε σχέση με το σημαντικότερο μέτρο σύγκρισης και τα υπόλοιπα και ένα άλλο το οποίο ήταν ενσωματωμένο στην πρόταση το τι θα κάνουμε για το καθεστώς ε, τρίτων ε, χωρών και βλέπω πως ε, η συγγήτρια τα αντιμετωπίζει αυτά επιτυχώς. Για τις επόμενες βλέπε, μέρες βλέπω κάτι ψηλοπράγματα αλλά να πω πως βρήκαμε νομίζω ένα συμβιβασμό που αφορά την κρισιμότητα των δικτών αναφοράς ε, και συμφωνώ επίσης με την αναλογικότητα μεταξύ κρίσιμων και μη δικτών αναφοράς Η δομή τώρα της πρότασης και των τροπολογιών είναι μια καλή φάση για να δούμε τι θα γίνει με τις τρίτες χώρες που ήταν ένα μικρό εμπόδιο στην αρχή. Τώρα έχουν μείνει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες και κάποια άλλα δευτερεύοντα ζητήματα. Εγώ θα ήθελα να δούμε τις τροπολογίες για την ε, νομική βεβαιότητα για τους χρήστες των δικτών αναφοράς και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για τις υποχρεωτικές συνεισφορές ε, τις τελευταίες ημέρες το θέμα των ε, δικτών αναφοράς για εμπορεύματα επίσης ε, άνοιξε. Ε, θα ήθελα να γίνουν και αυτοί οι δείκτες κάπως πιο ευρωστοί, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως το παράρτημα 1α κατά βάση ασχολείται με αυτούς οι οποίοι συνεισφέρουν και δεν υφίστανται κάποια ρύθμιση. Πρέπει λοιπόν να είναι και λειτουργικό το σύστημα. Τώρα, όσον αφορά το Συμβούλιο, εγώ στηρίζω τη δική μας την πρόταση απέναντι στο Συμβούλιο και την αναλογικότητα αυτή μεταξύ κρίσιμων και μη ε, δικτών αναφοράς. Αυτά και σας ευχαριστώ. Νομίζω και η κόρα και η ομάδα της κάνουν φανταστική δουλειά. Ευχαριστώ Λούντεκ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Άλβαρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κόρα για τα όσα έχει κάνει τους τελευταίους μήνες και να σας πω πως είναι πάρα πολλά, πολύ χρήσιμα για να πετύχουμε μια συμφωνία τουλάχιστον στο ιστορικό της Επιτροπή μας. Εάν αφήσω στην άκρη τις αρχικές μας παρατηρήσεις και αφήσω στην άκρη τις τροπολογίες και τους συμφιβασμούς που έχουμε μπροστά μας, θα πρέπει να εστιάσω καταρχήν στο γεγονός πως υπάρχει μεγάλη συμφωνία για τον ορισμό του ποιος είναι κρίσιμος δείκτης και πιστεύω πως η εισαγωγή κάποιων ποιοτικών ε, μεταβλητών ε, βελτιώνει τα πράγματα γιατί στην πρόταση της Κομισιόν έχουμε ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να έχουμε ορισμού οι οποίοι να συμπεριλαμβάνουν μόνο ποσοτικές μεταβλητές. Επίσης, ευρωπαϊκοί δείκτες. Αυτό επιτρέπουν κάποια κράτη-μέλη να ορίσουν ποιοι είναι οι δείκτες οι οποίοι για τους ίδιους είναι κρίσιμοι και αυτό σημαίνει πως για τους συγκεκριμένους χρειάζεται πιο αυστηρή νομοθεσία. Για το δεύτερο κεφάλαιο Πρέπει να σας πω πως η ομάδα των σοσιαλιστών δημοκρατών αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα. Το Συμβούλιο, όπως είπε και ο συνάδελφος από το ΕΛΚ, ακολουθεί μια προσέγγιση αναλογική μεταξύ των κρισίμων και μη κρισίμων δικτών. Και σε γενικές γραμμές πιστεύω πως είναι δυνατόν να αυξήσουμε αυτή την αναλογικότητα μεταξύ, μάλλον τη σχέση ε, μεταξύ κρισίμων και μη κρισίμων και αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς είναι να μελετήσουμε πιο βαθιά ποιοι είναι οι δείκτες και ποιες είναι οι απαιτήσει που θα θέλαμε να επιβάλλουμε ως μη κρισίμους. Και στο κεφάλαιο αυτό οπωσδήποτε να εισάγουμε και μία περιγραφή για το πώς θα αντιμετωπίζουμε τους μη κρίσιμους ε, δείκτες όταν μιλάμε για οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι εποπτευόμενοι, δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για εθελούσιες ε, συνεισφορές, γιατί για την περίπτωση των αγαθών ξέρετε πως δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή. Για να σας δώσω ε, μία άποψη για το τι πιστεύουμε εμείς για τους μη κρίσιμους δείκτες, η δική μας άποψη είναι πως θα πρέπει να δούμε πώς τις απαιτήσει που υπάρχουν για τους ε, οι δείκτες που, στους οποίους συνεισφέρουν ε, με εθελοντικό ε, τρόπο κάποιες οργανώσεις ή φορείς θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να αποτυπώσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια πώς θα γίνεται. Τώρα, για το σύστημα ισοδυναμίας, για την αναγνώριση δικτών, που έχουν ε, προετοιμάσει άλλα κράτη, να σας πω πως η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Γιατί δεν υπάρχει ισοδύναμη νομοθεσία στις δικές μας, στις μας, ε, στα δικά μας εσωτερικά δίκαια, οπότε καταλαβαίνει είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσουμε ως, ισοδύναμους, ως ισοδύναμη νομοθεσία από τρίτες χώρες. Πάντως πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί στους σημερινούς ε, συμβιβασμούς απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει κανείς δείκτες στους οποίους έχουν προετοιμάσει τρίτα κράτη τα οποία δεν καλύπτονται από διατάξεις περί ισοδυναμίας ειδικά όταν το σύστημα που χρειάζεται για την αναγνώριση δεν κρίνεται ως ισοδύναμο και αυτό για τους υποπτευόμενους ε, φορείς. Αν λοιπόν και αυτό με ανησυχεί. Αν απλώς απαγορεύσουμε αυτούς τους δείκτες για τους υποπτευόμενους φερείς, ε, τότε αυτό που ουσιαστικά κάνουμε είναι να ανοίξουμε μια πόρτα και να πούμε ότι οι υπόλοιπε επιχειρήσει, η υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία μπορούν να χρησιμοποιήσουν του δείκτε αυτού. Δηλαδή οι μη εποπτευόμενοι. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ρεαλιστική λύση. Δηλαδή αυτό το fair country regime που έχουμε και που βρίσκεται στο κείμενο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ένα ρεαλιστικό τρόπο για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό με αποτέλεσμα να το διευρύνουμε έτσι ώστε να καλύπτουμε όλους τους φορείς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους δείκτες και όχι μόνο τους εποπτευόμενους. Το εποπτικό πλαίσιο και ο ρόλος που θα έχει αυτό θα πρέπει να πιέζει προς μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, και των Ευρωπαϊκών ε, αρχών, γιατί όπως το Euribor ας πούμε επηρεάζει πάρα πολύ τα κράτη-μέλη, νομίζω πως θα πρέπει και εδώ να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία να παίξει ένα πιο συγκεκριμένο και πιο έντονο ρόλο και επαναλαμβάνω πάντα σε συνεργασία με την αρμόδια εθνική αρχή. Θα ήθελα να κλείσω ευχαριστώντας μια φορά ακόμα την κόρα ε, και την ομάδα της. Συνεργασήκαμε πάρα πολύ καλά και πρέπει να σου πω πως ο ορισμός του κρίσιμου δείκτη πιστεύω πως η εναλλακτική του Fair Country Regime θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις μη, τους μη εποπτευόμενους φορείς που μπορεί να αναλάβουν ε, και, και μάλιστα δίνοντας έναν πιο ορατό ρόλο στην, ε, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία αυτή και σχετικά με την ε, κατανομή μεταξύ κρισίμων και μη κρισίμων, νομίζω ότι θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε περισσότερο με τι υφιστάμενε υποχρεώσει και δεσμεύσει μα για να εξασφαλίσουμε πω αυτοί οι κρίσιμοι δείκτε ή αυτοί οι οποίοι ενδεχομένω θα γίνουν κρίσιμοι να έχουν ένα σφριγιλό πλαίσιο απαιτήσεων και για τους μη κρισίμους να βρούμε μια σταθερή σχέση για το σύνολο των δικτών έτσι ώστε ε, να καλύπτουμε και αυτούς οι οποίοι ε, είναι μέσα στο εθελούσιο σύστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ECR. Στη θέση της Κρίστιν Μπέρν μιλάει ο κύριος Λόντς. Ναι, η Κέι ζητάει συγγνώμη γιατί έχει αρρωστήσει. Θέλω να ευχαριστήσει την κυρία Φανιούν Χάιζεν για τη δουλειά που έκανε και την πάρα πολύ καλή συνεργασία και ειδικά για τις συμβιβαστικές προτάσεις. Ελπίζουμε λοιπόν έτσι να γίνει η ψηφοφορία ε, στην ώρα της στο Στρασβούργο. Τονίζει η ΚΕΙ πως ε, στις ε, προτάσεις της Κομισιόν δεν αναφέρεται και δεν ξεκαθαρίζεται το τι είναι ένα κρίσιμος δείκτης αναφοράς και δεν, αναφέρεται, και δεν καταλαβαίνουμε άρα τι θα καλύπτεται από τον ορισμό και τι όχι. Το γιατί επέλεξε η Κομισιόν τα 500 εκατομμύρια ευρώ ως το όριο για την κρισιμότητα και πώς θα υπολογίζεται αυτό. Και επίσης πώς μπορεί η Κομισιόν να την πάρουν σε σοβαρά όταν μιλάει για καλύτερη ρύθμιση όταν δεν μπορούν να μας δώσουν έναν κατάλογο του τι θα ρυθμίζει ε, η νέα αυτή ρύθμιση που προτείνουν. Ίσως λοιπόν μπορεί να τα απαντήσει αυτά η Κομισιόν αργότερα οι συμβιβαστικές προτάσεις της εισηγήτριας που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να κάνουν κάποιες ε, μη κρίσιμους δείκτες ε, κρίσιμους είναι, αν είναι συστημικά σημαντική, είναι κάτι το οποίο μπορεί να στηρίξει η ΚΕΙ, οπότε εδώ πέρα συμφωνεί μαζί σας η ΚΕΙ, κυρίως καθώς ο ορισμός ε, του κρίσιμου δεν είναι ορισμός. Επίσης η ΚΕΙ θα ήθελε να επαναλάβει το αίτημά της για την Κομισιόν για να φέρει μια, ε, έναν κατάλογο για το ποιοι δείκτες ε, είναι κρίσιμοι πάνω από αυτό το κατόφλι των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το άλλο βασικό ζήτημα ε, μοιάζει να είναι και δεν υπάρχει ακόμα στις συμβαστικές προτάσεις είναι κάτι το οποίο δεν ανέφερε μόνο η Κέι και το ECR, αλλά και τροπολογίες άλλων δύο πολιτικών ομάδων. Αυτό το οποίο σχετίζεται δηλαδή με τους δείκτες για εμπορεύματα, που δεν πρέπει να ρυθμίζονται σε αυτή την νομοθεσία, η οποία αφορά δείκτες αναφοράς ε, χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Νόημα της πρότασης είναι να υπάρξει κάποια ασφάλεια στο οικονομικό σύστημα και δεν μπορεί άρα να εφαρμοστεί σε οντότητες οι οποίες δεν, δεν υποπτεύονται και είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έχουμε δουλειά ακόμα. Με το να συμπεριληφθούν επίση και τα εμπορεύματα απλά δημιουργούμε την ψευδέστηση ότι έχουμε ρυθμίσει κάτι αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι αδύνατο να γίνει τα νομικά ζητήματα τα οποία δημιουργούν υποχρεώσεις ε, σε οντότητες είτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εκτός της δικαιοδοσίας ε, των υποπτικών αρχών είναι πάρα πολλά. Και η θεωρεί πως θα πρέπει να υπάρξει ένας ξεχωριστός κανονισμός για τα εμπορεύματα ο οποίος θα αναγνωρίζει το πώς λειτουργούν αυτές οι αγορές ε, και θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι καλή ιδέα να τα ανακατέψουμε αυτά. Ελήψη ε, αυτού. Οι δείκτες για τα εμπορεύματα καλύπτονται ήδη από την ε, οδηγία περί της ε, αγοράς και υπάρχουν άρα διοικητικές και ποινικέ κυρώσεις ε, και ελπίζει και ύπος και οι επόμενες ε, συναντήσεις και οδών θα έχουν μεγάλη συμμετοχή και θα αναφερθούν αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τη Μαρίζα από την ΚΟΥΕ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει τον λόγο. Όχι. Φίλιπ Λάμπερτς λοιπόν για τους πράσινους. Έχεις δίκιο ότι θα πρέπει να είναι να έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά ακούγοντας και παρατηρήσεις όπως αυτές της συναδέλφου ε, Κέι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να συγκρίνουμε ε, αντίθετα μεταξύ τους ε, πράγματα. Τα σχόλιά μου τώρα θα είναι περιορισμένα το γεγονός ότι προτείνεις ένα πιο ελαφρύ καθεστώς ε, για τους ε, μη κριτικούς δείκτες αναφοράς, μη κρίσιμους, ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό και συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν συμφωνούμε με τους συντηρητικούς. Είναι καλό να ε, μπαίνουν ε, και οι commodity benchmarks, αλλά ε, ο πιο σημαντικός δείκτης αναφοράς για τα, ο πιο σημαντικός commodity δείκτης αναφοράς είναι αυτός για τα πολύτιμα μέταλλα και ξέρουμε ότι εκεί θα έχουμε δυσκολίες. Εάν πρόκειται να εφαρμόσουμε κάτι θα πρέπει να είναι το ίδιο πάνω από ένα κατόφλι. Ε, υπάρχουν και δύο ορισμοί που λείπουν κατά την άποψή μας όσον αφορά δηλαδή ε, τον δίκτυο αναφοράς ε, της, των συναλλαγών και της ισοτιμίας και επίσης θα πρέπει να μας πείτε αν και κατά πόσον μπορείτε να στηρίξετε κάποιες τροπολογίες για θέματα ε, που δεν, έχετε που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αρχικό κείμενο. Επίσης, ε, ε, λείπει η έννοια του βασικού κινδύνου. Ε, ας πούμε ο Λίμπορ ε, χρησιμοποιείται για να καθορίζονται ε, ας πούμε τα μεταβλητά επιτόκια των ενυποθήκων στεγαστικών δανείων αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη ο βασικός κίνδυνος τα δύο πράγματα είναι ε, συνδεδεμένα, δηλαδή καθορισμός του βασικού κινδύνου αφενός και από την άλλη η σωστή χρήση των δικτών αναφοράς. Δηλαδή θα πρέπει να ε, είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει και η έννοια του βασικού κινδύνου, θα υπάρχει και η έννοια της σωστής χρήσης των δικτών αναφοράς. Θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια. Πιστεύω πάντως ότι οι δείκτες αναφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καταλήλως. Δεν πρέπει βέβαια να, δώσουμε εξαιρετικά συσταλτικέ ερμηνείε των όρων, αλλά παρόλα αυτά να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά το κατά πόσο είναι κρίσιμοι ή όχι κάποιοι δείκτες. Είπαμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κριτήρια ποσοτικά και ποιοτικά ε, για τον καθορισμό των, της χρησιμότητας των δικτών. Ε, πιστεύουμε ότι 100 εκατομμύρια θα πρέπει να είναι το όριο Εκατό δις θα πρέπει να είναι το, όριο. Ε, και εδώ πρέπει να πω ότι η συγγέντρια της Άλντε μας εκπλήσει λίγο διότι ε, αφήνει τον ορισμό του, του βαθμού της κρισιμότητας των δικτών αναφοράς στις εθνικές αρχές. Αλλά εάν κανείς αφήσει αυτού του είδους την αξιολόγηση στους εθνικούς επόπτες, τότε ε, διατρέχει τον κίνδυνο να έχει τελείως διαφορετικά πρότυπα, άρα ε, και στρέβλωση της αγοράς. Θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό και να δούμε και πώς ε, ε, ήταν η πρόταση της Κομισιόν η οποία έλεγε ότι θα πρέπει ο ορισμός ε, να αποφασίζεται και να εφαρμόζεται σε ενωσιακό επίπεδο. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε στον κανονισμό βέβαια, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει σαφώς να αναφερθεί ότι κάτι, μια τέτοια απόφαση δεν μπορεί να αφαιθεί στους εθνικούς επόπτες. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι συμβιβασμοί που είδαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, ε, καλούμε το, την ΕΣΜΑ να παίξει σημαντικό ρόλο. Ξέρουμε ότι πολλοί δείκτες ε, αναφοράς παράγονται, ας πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, και Ξέρουμε ότι ακριβώς στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν γίνει οι χειρότερες ε, καταχρήσεις ε, και παραβιάσεις. Επομένως, ε, αυτό είναι γνωστό. Πιστεύουμε ότι όσον αφορά τους κρίσιμους δείκτες ε, αναφοράς ε, ο, ο κανόνας θα είναι ότι θα πρέπει να αποφασίζονται σε ενωσιακό επίπεδο. Ξέρουμε ότι για χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο ε, και σε αυτές τις περιπτώσεις ενδεχομένως μπορούμε να ζητήσουμε από την ΕΣΜΑ να πάρει θέση αντί για το κράτος. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι κανονικά ο, ο, κανόνας λέει ότι η ΕΣΜΑ ε, ε, ε, παίρνει τις αποφάσεις και είναι αυτή που εποπτεύει αλλά μπορεί ε, να ε, μετακυλήσει ας πούμε κάποια ευθύνη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και σε περίπτωση που κάποια στιγμή ε, θεωρεί με σωστά επιχειρήματα ε, ότι δεν γίνεται καλά ε, η δουλειά σε εθνικό επίπεδο, τότε να αποσύρει αυτήν την μετακύληση της αρμοδιότητας. Γιατί ξέρουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν γίνει πολλές καταχρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι εάν η ΕΣΜΑ διαπιστώσει ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ε, ε, εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο και την ανάληψη αρμοδιοτήτων σε εθνικό επίπεδο, τότε να είναι σε θέση να ξαναείχει το δικαίωμα να ξαναπάρει πίσω την ε, δυνατότητα εποπτείας. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι οι χώρες δεν κάνουν καλή δουλειά ή δεν μπορούν να κάνουν καλή δουλειά, αλλήμωνο αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να διατηρήσουμε το δικαίωμα εάν ε, προκύψει ανάγκη και κατά περίπτωση να μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτή τη δυνατότητα από τις χώρες ε, Θα, τα δου, θα πρέπει να δούμε και τις ε, συμβαστικές λύσεις στις οποίες έχουμε φτάσει σε προηγούμενα κείμενα και προηγούμενα επίπεδα αλλά επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να παραμείνει η δυνατότητα της ε, ενωσιακής αρχής να ξαναπάρει την ε, αρμοδιότητα εάν δει καταχρήσεις. Όσον αφορά τώρα τα ισοδύναμα, ισοδύναμες απαιτήσει για τρίτες χώρες, ε, θα ήταν καλό ε, εάν οι σκιώδεις εισηγητές, ε, οι ε, μπορούσαν να συμφωνήσουν σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να λέει ότι θα πρέπει να προσέχουμε έτσι ώστε οι τρίτες χώρες να μην παρουσιάζουν χαρακτηριστικά φορολογικών παραδείσων και επομένως θα πρέπει τα ισοδύναμα να καθορίζονται πολύ αυστηρά έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, οι τρίτες αυτές χώρες να λειτουργούν σαν φορολογική παράδειση. Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια ευρεία συμφωνία όσον αφορά το θέμα αυτό και να πω στους συναδέλφους του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν είναι εδώ, που είναι απόντες, ότι αναγνωρίζουμε ότι έχει ε, γίνει μεγάλη πρόοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο που αφορά την κύρια χρηματοπιστωτική αγορά ε, της Ευρώπης ε, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν ξανά προβλήματα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν έναυσμα για πολύ μεγάλη δυσκολία. Ευχαριστώ Φίλιπ. Εξακολουθώ να μην βλέπω κανέναν από την ΚΟΕ. Κοιτάω και το χρόνο, οπότε ανοίγω τη γενική συζήτηση. Ε, θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος να ε, πει κάτι. Αν δεν θέλει κανείς να πει τίποτα, να δώσω ξανά το λόγο απευθεία στην κόρα. Α, η Κομισιόν, με συγχωρείτε. Πήγανε τα πράγματα πολύ γρήγορα γι' αυτό. Ε, ευχαριστώ που ήρθατε και αναμένουμε να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά από τη συζήτηση αυτή έχω κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα το ότι η Κομισιόν παρουσίασε αυτή την πρόταση για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στους δείκτες αναφοράς μέσω της αξιοπιστίας των δικτών. Κοιτάξτε, εμείς ακολουθήσαμε τις αρχές της ΙΟΣΚΑ για να δούμε την ε, ποιότητα των δεδομένων, τον έλεγχο, την διακυβέρνηση, να υπάρχουν επαρκή δεδομένα, όπως είπα, και βεβαίως να διασφαλίσουμε πως υπάρχει και επαρκής προστασία των καταναλωτών. Θα ήθελα εδώ πέρα να πω πως χτες η ΕΣΜΑ δημοσίευσε μια έκθεση για την ε, εφαρμογή των αρχών της ΕΣΚΟ. Θα το βρείτε στη σελίδα της. Και η έκθεση δεν είναι τόσο καλή όσον αφορά την ε, συμμόρφωση όλων των παρόχων δικτών αναφοράς γιατί είδαμε σε κάποιες ε, τροπολογίες που κατατέθηκαν πως ε, οι μη κρίσιμοι δείκτες δεν θα υπόκεινται στους δείκτες, στους, στις αρχές της ΑΙΟΣΚΟ. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουν ε, οι Ευρωπαίοι πάροχοι τέτοιων δικτών σε σχέση με τις αρχές της ΑΙΟΣΚΟ. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω εδώ πέρα τους δείκτες για τα εμπορεύματα, οι οποίοι επίσης ε, καλύπτονται από τις αρχές της ΑΙΟΣΚΟ, οπότε ε, θα πρέπει να υπάρχει και εδώ πέρα στη βαρύ διακυβέρνηση και συστήματα ελέγχου για να συντάσσονται αυτοί οι δείκτες και βεβαίω πράγματι πρέπει να ισχύσει αναλογικότητα σε σχέση με το πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι αρχές στους διάφορους δείκτες αναφοράς αλλά οι γενικές αρχές θα πρέπει να διατηρηθούν για όλους τους τύπους δικτών. Δεν βλέπουμε τώρα κάποιο λόγο για να ξεκινήσουμε την συζήτηση ξανά όταν η ΑΙΟΣΚΟ έχει αναγνωρίσει στην εφαρμογή των αρχών πως αυτά ισχύουν και για τους δείκτες εμπορευμάτων. Με τα δύο άλλα πράγματα, το πρώτο για τον καθορισμό των κρισίμων. Εμείς, ορίσαμε, εμείς χρησιμοποίησαμε τον ορισμό του κρίσιμου απλά για να υπάρξει η σύσταση ενός σώματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βεβαίως να ε, υπάρχει και η δυνατότητα σε εθνικό επίπεδο να υπάρχει η συμμετοχή σε αυτά τα σώματα. Δεν υπάρχει επιπλέον αναλογικότητα. Οπότε αποφασίσαμε να βάλουμε έναν ορισμό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ στενός και περιορισμένος και αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι πως δεν μπορούμε σήμερα να δώσουμε κάποιον κατάλογο, δεν, έχουμε τα δεδομένα, δεν έχω τα δεδομένα εδώ πέρα τώρα, αλλά το σκεπτικό μας ήταν να καλύψουμε μόνο ελάχιστους δείκτες ε, επιτοκίων, γιατί οι οντότητες αυτές θα έπρεπε να έχουν κάποια υποπτία ε, Euribor δηλαδή, Libor, Σάιμπορ και ίσως ε, άλλος ένας, αλλά όχι πολύ. Οπότε, ε, λάβετε το αυτό υπόψη στη συζήτησή σας. Μετά το ζήτημα των τρίτων χωρών, να πω κάποια πράγματα. Γνωρίζουμε το ότι η ισοδυναμία από μόνη της δεν λειτουργεί. Το προτείνουμε γιατί όταν συντάχθηκαν οι αρχές ε, ΑΙΟΣΚΟ υπήρχε μια πρόταση που έλεγε ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη να τις εφαρμόσουμε κτλ. Και μετά από 1,5 χρόνο βλέπουμε πως αυτό δεν συμβαίνει σε πάρα πολλές ε, δικαιοδοσίες και για το λόγο αυτό θα θέλαμε να δούμε κάποιες άλλες ε, λύσεις για να βρεθεί ένας τρόπος για να χρησιμοποιηθούν οι δείκτες τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και πάλι αρκεί να είναι στιβαροί και αξιόπιστοι και να δημιουργούν ίσους όρους ανταγωνισμού. Σας ευχαριστώ κυρία Φερνάντες. Τον λόγο έχει η κυρία Νιουερχόιζεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα ενθαρρυντικά του σχόλια. Καταγράφω πως έχουμε ακόμα εκκρεμότητες που πρέπει να δουλέψουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντίδρασή τους. Θέλω να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Οπότε, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, ας συναντηθούμε με τους σκιώδεις και ας συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για το συμβιβασμό. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστούμε κόρα. Να πω επίσης ε, πώς θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 9 Μαρτίου και στην Ολομέλεια, στην δεύτερη Ολομέλεια του Μαρτίου. Περνάμε λοιπόν τώρα απευθείας, παρά το ότι είμαστε και λίγο πιο νωρίς. Για να μην κάνουμε διάλειμμα, περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης συστάσεις ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη ελλανδική ε, Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων TTIP. Κόρα, για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, για να μην ε, έχουμε προβλήματα, 9 Μαρτίου είχαμε πει να ψηφίσουμε, όχι 2 Μαρτίου. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση. Οπότε, περνάμε στο Σημείο 5. Δίνω τον λόγο στον Γέπε Κόφοντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω πως ε, είναι πιο νωρίς από ό,τι είχε προβλεφθεί στην ημερήσια διάταξη ε, το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι θα κάνουμε μια καλή συζήτηση. Καταρχήν, ευχαριστώ που δίνει την ευκαιρία αυτή να απευθυνθώ στην Επιτροπή. Ε, Τώρα, για την εντολή που έχουμε και για τα επίσημα κριτήρια για την γνωμοδότηση. Ξέρετε πως πολλές επιτροπές του Κοινοβουλίου στο δικό τους κλάδο κάνουν μια αντίστοιχη γνωμοδότηση. Θα ήθελα να έχουμε εκτός της εντολής της ΕΚΟ να προσθέσει και κάποια άλλα σημεία. Αλλά ξέρετε πως περιοριζόμαστε στο ε, μέγεθος των όσων μπορούμε εμείς να εκφράσουμε. Να σας πω πως για την Ευρώπη και για τις ΗΠΑ και για τη συμφωνία TTIP Πρέπει να θα οδηγηθούμε στη μεγαλύτερη διμερή επενδυτική συμφωνία και θα αποτελέσει ενδεχομένω και το χρυσό κανόνα για τι εμπορικέ επενδύσει και τι σχετικέ συμφωνίε. Βασίζεται στη διαφάνεια, στο κράτο δικαίου και νομίζω θα αποτελεί υπόδειγμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να υποεκτιμήσουμε, ούτε είναι υπερβολή από μένα να υπογραμμίσω μια φορά ακόμα πόσο σημαντική είναι η γεωπολιτική διάσταση αυτή τη συμφωνία εμπόριο, θέσει απασχόληση οικονομικά αλλά και γεωπολιτική συνεργασία με, τα, με ΣΥΠΑ. Τώρα, τι πιστεύουμε στην ΕΚΟΝ για την TTIP. Ο ανταγωνισμό, οι κρατικέ επιδοτήσει, οι πρόσβαση αγορά, οι κρατικέ επιχειρήσει και οι χρησιμοποιητικές επιχειρήσεις είναι σημαντικά για μα. Κάποια από τα θέματα που έχω συμπεριλάβει στη γνωμοδότηση έχουν ε, σχέσει και με τα όσα θα πούν οι άλλε επιτροπέ. Όμω είναι απαραίτητο αυτό. Γιατί ο ανταγωνισμό είναι το δικό μα, ε, αν θέλετε, χωράφι και είμαι εδώ για να ακούσω και τις δικές σας απόψεις και να είμαστε σίγουροι πως οι γνωμοδοτήσεις της, στην ΕΚΟΝ και η προσφορά μας στην ε, απόφαση της ΙΝΤΑ θα καλύπτουν όλες τις δικές σας απόψεις. Στην πρώτη παράγραφο λέω πως η συμφωνία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε, χαμηλότερα, σε, χαμηλότερους, σε χαμηλότερο επίπεδο προστασίας. Δηλαδή θα πρέπει τα πρότυπα που ακολουθούμε στο περιβάλλον, και νομοθεσία να ακολουθούν αυτά τα οποία εμείς πρεσβεύουμε. Δεν έχω χρόνο να μπω με λεπτομέρειες όλες τις παραγράφους. Θα ήθελα λοιπόν να εστιάσω σε κάποιες οι οποίες έχουν συζητηθεί περισσότερο στις διμερείς συναντήσεις μας. Αν δείτε την παράγραφο Δέλτα, θα δείτε πως μιλά για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Είναι μία από τις δικές μας αρμοδιότητες εδώ στη δική μας Επιτροπή. Γίνονται αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις για το θέμα εκτός ε, του χώρου της TTIP και ανεξάρτητα από που γίνονται οι διαπραγματεύσεις, εγώ πιστεύω πως ο στόχος μας είναι καταρχήν πολύ ε, υψηλό επίπεδο προστασίας για το περιβάλλον, για τις εργασιακές σχέσεις και για την προστασία της υγείας και της υγιεινής. Αν λοιπόν θα πρέπει να συγκλίνουμε προς τα πάνω, τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να ορίσουμε όλα τα θέματα έτσι ώστε να αποφύγουμε την διασπορά ε, οποιασδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική χρηματοπιστωτική κρίση. Στην παράγραφο I μιλάω για το ISDS, δηλαδή ε, για την διακανονισμό διαφορών σε θέματα επενδύσεων. Και σε σχέση με την εντολή της ΕΚΟΝ, να σας πω πως το θέμα το δικό μας είναι πώς θα επιλύονται αυτές οι διαφωνίες που προκύπτουν από την πρόσβαση στην αγορά και όπως επίσης από κάποια θέματα ανταγωνισμού. Πιστεύω πως τα εθνικά δικαστήρια και τα συστήματα ε, ε, τα εθνικά θα πρέπει να ακολουθούν την εξή αρχή. Πρώτον, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ βασίζονται σε δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και την διαφάνεια. Άρα λοιπόν θεωρούν πως η έννοια της αυτόματης χρήσης μιας, ε, ενός μη κρατικού μηχανισμού είναι προβληματικός. Όμως, μπορεί να προκύψουν κάποιες περιστάσεις, κατά τις οποίες χρειάζεται μια τελείως αμερόληπτη ε, αξιολόγηση. Για παράδειγμα, εάν μια, μια υπόθεση ε, έχει πάει στα δικαστήρια και εκεί εκρεμεί για χρόνια. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να έχουμε αυτή τη δυνατότητα ε, ένας δηλαδή μηχανισμός επιδιαιτησίας μη κρατικός. Για τη διαφάνεια, πώς μπορούμε να το εξασφαλίσουμε αυτό με μη κρατικούς μηχανισμούς. Μία από τις σκέψεις που έκανα, γιατί σκέφτομαι πολύ για τα θέματα της διαφάνειας, είναι αυτός ο μηχανισμός διαιτησίας να μπορεί να χρησιμοποιεί ήδη τους υπάρχοντες, δηλαδή αυτοί που υπάρχουν από ε, την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπορικό Δίκαιο, Δηλαδή, ότι τα έγγραφα είναι προσβάσιμα και είναι δημόσια και πώς ε, επιλέγουμε τους ε, διαιτητές κτλ. Η τίτη πολύ συχνά αναφέρεται ως ο χρυσούς κανόνας για τις μελλοντικές ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Οπότε, εάν εμεί εντάξουμε ένα τέτοιο είδου μηχανισμό, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί αν έχουμε τέτοια συμφωνία, πώ θα έχουμε ένα μη κρατικό μηχανισμό επίλυση διαφορών, αν οι χώρε με τι οποίε έχουμε συνάψει συμφωνία δεν βασίζονται στι δημοκρατικέ αρχέ και στο κράτο δικαίου. Θα δώσω τώρα το λόγο Στου σκιώδεις ε, εισηγητές και πρέπει να σας πω πως περιμένουμε ανυπομονησία τις δικές σας ιδέες και τα δικά σας σχόλια έτσι ώστε η συνεισφορά τη ΕΚΟΝ στην ε, έκθεση της ΙΝΤΑ για την TTIP ακόμα πιο ε, αποφασιστική. Ευχαριστώ Γέπε. Μια που η Ντανούτα Χίμπνερ ισχυώδης για το ΕΛΚ δεν είναι εδώ, έχουμε έναν άλλον συνάδελφο όμως ο οποίος θα μιλήσει για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ντανούτα Χούμπνερ ε, δεν είναι εδώ σήμερα. Και ε, μου ζήτησε να μεταφέρω τα σχόλιά της ε, για την έκθεση του κυρίου Γκόφερ και να τον ευχαριστήσει για τη δουλειά που έχει κάνει. Έχει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις Πρώτα απ' όλα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και μετά βέβαια να δούμε το ζήτημα του ISDS και Τέλος, οι παρατηρήσεις της εστιάζονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πόρος πρέπει να βελτιωθεί ο ρόλος τους εντός των διαπραγματεύσεων TTIP και ελπίζουμε να καταθέσει κάποιες τροπολογίες για τις ε, υπηρεσίες, ε, τις χρηματοπιστωτικές όπως είπε ο εισηγητής. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις στον τομέα αυτών με τρόπο θετικό και βεβαίως λαμβάνοντας είναι το ότι έχει επιτευχθεί σήμερα και στις δύο όχθες του Ατλαντικού και κατά την άποψη της Ντανούτας οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διμερείς διαβουλεύσεις ε, πριν ε, ενεργοποιηθούν νέα νομοθετήματα. Θεωρεί λοιπόν πως θα πρέπει να υπάρξουν έντονες διμερείς συζητήσεις πριν υπάρξει νέα νομοθεσία δεύτερον για το θέμα της ε, διαφάνειας ε, ε, πρέπει να υπάρξει ειδικά στις διμερείς συνομιλίες και τέλος να υπάρξει λογοδοσία ερετών σωμάτων όπως και το Κοινοβούλιο για να υπάρξει και μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις και το STS θεωρεί πως η Κομισιόν πρέπει να εξετάσει την εισαγωγή ενός νέου μηχανισμού επίλυσης επενδυτικών διαφορών υπό την TTIP ε, μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα αντικαταστήσει τις διμερείς ε, επενδυτικές υφιστάμενες συνθήκες με τις ΙΠΑ. Και βεβαίως οποιοδήποτε τέτοιος μηχανισμός πρέπει να είναι διαφανής και να ελέγχεται με βάση δημοκρατικές αρχές ε, και να υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς ε, και μια δυνατότητα προσφυγής. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διαιτησία για να αποφεύγονται ε, συγκρούσεις και να μειωθεί το κόστος για να έχουν πρόσβαση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι το οποίο αξίζει επίσης να δούμε είναι πώς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής οι επενδυτές εντός του εγχώριου δικαστικού συστήματος. Θα πρέπει βεβαίω να δούμε και το τι γίνεται στο πλαίσιο του ISDS, να υπάρχει η δυνατότητα δηλαδή να προσφύγει κάποιος εκεί πριν πάει στα εγχώρια δικαστήρια. Τέλος, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κύριε Πρόεδρε, δεδομένου του ότι η TTIP θα ωφελήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο από τις μεγάλες, έτσι θέλουμε τουλάχιστον, θα πρέπει να απλοποιηθούν τελωνιακές διαδικασίες ε, και να ε, μετατραπούν οι διάφορες προδιαγραφές των προϊόντων και θα έχουμε την πρώτη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου που θα έχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα πρέπει άρα να κωδικοποιηθεί η φυστάμενη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υπάρχουν πληροφορίες σε κάποια site όπου και ευρωπαϊκές και αμερικανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να βλέπουν τους δασμούς, τις τελωνιακές διαδικασίες και όλους τους σχετικούς κανονισμούς σε ομοσπονδιακό και τοπικό επίπεδο. Η κυρία Χούμπνερ θεωρεί πως το βάρος της μικρομεσαίας επιχειρήσης, το ότι θα έχουν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο και το να φτιάξουμε ένα site είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο. Αναμένει λοιπόν την συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστούμε για το ECR Σανταλούτς. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούμε και διμερώς και να σχολιάσουμε το φάκελο. Οπότε με χαρά θα συνεργαστώ και μελλοντικά μαζί σας και βέβαια είμαι και αναπληρωτής στην ίντα οπότε καταλαβαίνετε ότι ο φάκελος τους με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Με την έκθεση αυτή λέμε πως θέλουμε μια φιλόδοξη συμφωνία με σωτιστήτη με πρόθεση της οικονομίας και στις δύο όχθες του Ατλαντικού, γιατί πολλοί λένε ότι οι ελεύθερες συναλλαγές ε, είναι πολύ καλή για την απασχόληση και την οικονομία, λίγο καλή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά κανείς δεν μιλά για το πόσο θετικό θα είναι για τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Γιατί αν είναι φθηνότερα τα αγαθά που θα αγοράζουν και καλής ποιότητας, τότε πραγματικά θα ευνοηθούν. Έτσι θα αυξηθεί και η ζήτηση για τις, χώρε υπηρεσίες και αυτό θα φέρει περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Τώρα για την έκθεση έχω πέντε σύντομες παρατηρήσεις. Όπως είπα προηγουμένως, βλέπω πως η έκθεση ε, εστιάζει περισσότερο στη θέμα του προστατευτισμού Νομίζω ότι θα πρέπει εμείς και τον ευρωπαϊκό προστατευσιμό να τον ξεπεράσουμε ε, γιατί πλήττει τους ευρωπαίους καταναλωτές. Επίσης, χρειάζεται να προωθήσουμε την ενισχυμένη συνεργασία και η γνωμοδότηση ξεκινά από τη σύγκληση. Να κάνουμε λοιπόν μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Τρίτον, φορολογική πολιτική. Κατά τη γνώμη μας δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το θέμα αυτό στην TTIP. αλλά θα πρέπει να δούμε ίσως το θέμα της πολιτικής ανταγωνισμού. Γιατί έχουμε κάποιες διατάξεις που ενδεχομένως μπορεί να καλύπτουν τις συγχωνεύσεις και τη δημιουργία τραστ, τις επιδοτήσεις σε κρατικές επιχειρήσεις κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα με τον ανταγωνισμό και καλό θα ήταν να το θίξουμε και στην έκθεση. Τέταρτον, συμμερίζουμε απόλυτα την άποψη του ε, εισηγητή πως χρειαζόμαστε το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας. Εδώ δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Και τέλος, συμφωνώ με τον εισηγητή, θα πρέπει να δούμε ένα καλύτερο τρόπο να προστατευτούν οι επενδύσεις και αυτό προστατεύοντας παράλληλα την νομοθετική μας, τα νομοθετικά μας δικαιώματα, γιατί αυτό θα επιτρέψει σε επενδυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, τύχουν μιας ε, δίκαιης συμπεριφοράς, αλλά ίσως για το θέμα αυτό το χρυσό δισκοπότηρο δεν θα το βρούμε ακόμα σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, στο μέλλον σίγουρα θα έχουμε και κάποιες καινούργιες ιδέες για να εμπλουτίσουμε το θέμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Άλντε Ραμόν Τρεμόζα για την Κούε Μακάρθη και τη Μαρίζα. Βλέπω, οπότε θα δώσω τον λόγο στους ε, πράσινους ε, στον ε, Μιχέλ Ρεμόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για εμάς τι είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν τους επόμενους μήνες. Για την έκθεση ΕΚΟΝ, της ΕΚΟΝ ε, έχουμε να παρατηρήσουμε το εξής. Η περαιτέρω απορρίθμιση των χρηματαγορών δεν είναι πλέον επιλογή για εμάς και δεν μπορούμε να την στηρίξουμε. Και θα θέλαμε η έκθεση της ε, Οικονομικής Επιτροπής να προωθεί την περαιτέρω και την καλύτερη ρύθμιση και όχι την απορρίθμιση. Και μετά ζητείτε εδώ πέρα να μπουν κάποιες προδιαγραφές ειδικά αυτές που, που ισχύουν στις ΗΠΑ. Κοίταξε, κάποιες από τις προτάσεις μας ε, θα πάνε προς την κατεύθυνση καλύτερης ρύθμισης ε, των χρηματαγορών και των αγορών των ασφαλιών. Αυτό ισχύει ειδικά για την ρυθμιστική συνεργασία. Θεωρώ πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ πέρα πρέπει να είναι σαφώς υπέρ. Και θα πρέπει η ρυθμιστική εποπτεία να βρίσκεται 100% στα χέρια των κοινοβουλίων. Έχουμε δικαίωμα στη ρύθμιση και δεν πρέπει να εξασθενήσει αυτό. Ένα άλλο σημαντικό είναι επίσης οι δημόσιες προμήθειες. Καθώς υπάρχει εδώ πέρα η δυνατότητα να σταματήσει η φυστάμενη κατάσταση, αυτό πάει προς τη τελείως λάθος κατεύθυνση. Θα πρέπει οι προμήθειες να γίνονται τοπικά με, κοινωνική και οικολογική υπευθυνότητα. Και το τελευταίο, εννοείται πως θεωρούμε πως η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να σταθεί ξεκάθαρα κατά των μέτρων προστασίας των επενδυτών του ISDS. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ρεμόν. Για το EFTD ε, πάλι δεν βλέπω κανέναν. Έρχεται όμως ο συνάδελφος από τους φιλελεύθερους. Δεν ε, έχει ιδέα τι τον περιμένει. Αλλά ούτε αυτός μάλλον αντικαθιστά τον Ραμόν Τρεμόζα ή όχι. Δεν ξέρω ε, παίρνετε αμέσως τον ε, λόγο. Ε, έπρεπε να... Ξεκινήσατε ήδη τη συζήτηση για το TTIP. Α, ζητώ συγγνώμη, ήμουν στο γραφείο μου και ε, έλεγα ότι θα ξεκινήσει σε πέντε λεπτά. Ναι, ναι, συγγνώμη, προχωρήσαμε λίγο γρήγορα. Με συγχωρείτε και εμένα, λέει ο Uh, Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τον συντάκτη της γνωμοδότησης, τον κύριο Κόφορτ. Διότι πάντα ήταν ανοιχτή η πόρτα του και είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Ε, πρέπει η συμφωνία να είναι όσο ευρύτερη γίνεται σε αυτό το θέμα. με ικανοποιεί το κείμενο που μας έχει υποβάλει. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε όχι ακριβώς αλλαγές, αλλά ίσως να χρησιμοποιήσουμε διαφορετική διατύπωση. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά συμφωνώ απολύτως με τα κεντρικά του σημεία. Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση που είναι υποβοηθητική των επιχειρήσεων. Πρέπει να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, γιατί αν τώρα πούμε όχι καθαρό ε, σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, ποιε θα είναι οι ευκαιρίες για την Ευρώπη, ποια είναι η εναλλακτική. Μεγάλες πολυεθνικές ε, από την ε, Ευρώπη δρούν στην, είναι παρούσες στις ΗΠΑ και ισχύει και το αντίστοιχο εδώ και πολλά χρόνια μάλιστα. Εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε για δασμούς, μπορούμε να μιλήσουμε ε, για ε, τελωνιακά, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα σωρό πράγματα τα οποία μπλοκάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και πολλά χρήματα, πολλοί πόροι χρησιμοποιούνται, ε, δαπανώνται έτσι ώστε να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία και να ξεπεραστούν όλα αυτά τα προσκόμματα και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία, όπως άλλωστε λέει και η γνωμοδότηση. Χρειαζόμαστε επίσης διαφάνεια, χρειαζόμαστε ε, ε, σαφή τοποθέτηση για το κατά πόσο θα περιλαμβάνονται ή όχι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα υπάρχει διαφάνεια στη ροή κεφαλαίων ένθεν κακήθεν. Και βεβαίως να να διαβεβαιώσουμε ότι να εγγυηθούμε ότι ε, δεν θα υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού ή φορολογική στρέβλωση για τις εταιρείες ε, ανάλογα με το ε, αν δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες ή στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα διατύπωνα ίσως διαφορετικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, έχουμε παράδοση υπέρ της δημόσιας ε, υπηρεσίας ή των δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό μπορεί κανείς να το κατανοήσει όπως θέλει. Θα μπορούσε να ε, σημαίνει αυτό ότι θέλουμε μονοπόλια εις βάρος του ιδιωτικού τομέα. Αυτό δεν μπορούσε να διατυπωθεί λίγο διαφορετικά. Ε, και βεβαίως θέλουμε μια διατύπωση η οποία ε, δεν θα, ε, θα δημιουργεί κανένα πρόβλημα στο κράτος ε, κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, αυτό που διαπιστώνω, μάλλον να το πω διαφορετικά, Μπορώ να σας πω ότι έγινε στην Αργεντινή πριν από δύο χρόνια. Ε, υπήρχε η, ισπανική εταιρεία ε, Repsol, ε, η οποία, την οποία έδιωξε στην ουσία η κυβέρνηση κρατικοποιώντας την εταιρεία. Νομίζω ότι εάν δεν υπήρχαν διεθνείς κανόνες τα προβλήματα θα ήταν ε, πολύ περισσότερα. Without any compensations. Because... Ε, βεβαίως ε, στην προκείμενη περίπτωση η κυβέρνηση της Αργεντινής δεν δίμευσε το 100% της ε, Ρεψόλ, ε, γιατί ήξερε ότι διαφορετικά θα βρισκόταν αντιμέτωποι με τους ε, διεθνείς κανόνες. Αλλά θα πρέπει να, λάβουμε, να ληφθούν υπόψη και οι εθνικές νομοθεσίες, αλλά ταυτόχρονα είτε να δημιουργηθούν είτε να διατηρηθούν κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Να δούμε πώς μπορούμε δηλαδή να έχουμε ένα συνδυασμό όλων αυτών των στοιχείων. Όσον αφορά το ESDS, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ε, ξέρουμε και ότι στην Λατινική Αμερική είναι καλύτερη, στην Αμερική συγγνώμη, είναι η καλύτερη δικηγόρη ε, και επομένως